απολογίες. Τώρα, με βάση την ημερήσια διάταξη, έχουμε την ερώτηση προς το Συμβούλιο ε, σε σχέση με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων και έχουν πρώτα το λόγο η κυρία Χάουταλα για τρία λεπτά. Κάνω Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η Σουηδική Προεδρία έθιξε το θέμα της οικοδόμησης δημοκρατίας ως ένα τμήμα των προτεραιοτήτων της στις εξωτερικές δράσεις. Ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέλω να απογραμμίσω ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα υπάρχουν ε, διάφορες ερμηνείες στις δημοκρατίες όπου με τον ε, ένα ή τον άλλο τρόπο εμφανίζονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ορίζοντας τη δημοκρατία το 2005 τα Ηνωμένα Έθνη ε, παρέθεσαν την ελευθερία, το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και πάρα πολλά άλλα στοιχεία ως βασικά συστατικά της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως σας είπα είναι αναπόσπαστο τμήμα της δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εργαλειοθήκη της ας την πούμε έχει πάρα πολλά εργαλεία που στηρίζουν τη δημοκρατία, την ε, χρηματοδοτική πολιτική και πάρα πολλά άλλα. Ε, διεξάγουμε διάλογο με άλλες χώρες, έχουμε ε, στοιχεία χρηματοδότησης και η παρατήρηση των εκλογών είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα δική μας, όπως και το τι κάνουμε στα διεθνή φόρουμ. Υπάρχουν όμως καταστάσεις όπου είναι κανείς αναγκασμένος να εξετάσει και τις αρνητικές πτυχές της δημοκρατίας. Και εδώ ε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Υπουργού στο ότι ε, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πρόκειται να συζητήσει για την άρση του ε, εμπορίου όπλων με το Ουσμπεκιστάν. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι λάθος μήνυμα, διότι το Ουσμπεκιστάν αγνόησε τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας. Η διεθνής κοινότης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν μία σε βάθος ε, έρευνα αυτών των ε, τραγικών ε, γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Αντιτζάν όμως το Ουσμπεκιστάν δεν ανταποκρίθηκε. Γι' αυτό λοιπόν δεν κατανοώ γιατί θεωρείτε ότι έχει φτάσει η χρονική στιγμή για να άρουμε το εμπάργκο όπλων. Βέβαια η δημοκρατία δεν είναι εξαγώγημο προϊόν και δεν μπορεί κανείς να φυτεύσει τη δημοκρατία σε μια άλλη χώρα. Γι' αυτό το λόγο η κοινωνία των πολιτών καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η δημοκρατία ευδοκιμεί ξεκινώντας από τη βάση. Ε, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η Ρωσία είναι δικός μας εταίρος, ο οποίος συστηματικά αρνείται να επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών αλλά και ε, στις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις να έχουν πρόσβαση στο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα εξάλλου να πω ότι η οικοδόμηση της δημοκρατίας θα πρέπει να αποτελεί ε, πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική κέπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δηλαδή μεγαλύτερη χρηματοδότηση Επίσης ε, να ε, βελτιώσουμε και τα εργαλεία για την ε, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λόγο έχει η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αλμπερτίνη, κυρία Αντζελή για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα. Είναι η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που επιτρέπει να αναγνωριστεί ένα καθεστώς ως δημοκρατικό. Θα πρέπει λοιπόν να χαρούμε που τον Μάιο το Συμβούλιο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πιο συνεκτική προσέγγιση για την δημοκρατική ε, διακυβέρνηση. Αλλά τα μέτρα υπήρξαν μέχρι τώρα ανεπαρκή. Η ε, σύγκρουση ε, η Ισραηλο-Παλαιστινιακή είναι ένα κατάφορο παράδειγμα, ενώ η αποστολή για την παρατήρηση των εκλογών των Παλαιστινιακών του 2006 είχε αναγνωρίσει την ομιμότητα των αποτελεσμάτων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα κράτη-μέλη μποϊκόταραν την κυβέρνηση που προήλθε από τις εκλογές την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και Πού βρίσκεται η συνεκτικότητα και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι ίδιες οι αποφάσεις της είναι αντίθετες προς τις αρχές που διακηρύσει. Και τι να πούμε για ορισμένα κρατημέλη ε, που δεν υποστηρίζουν την έκθεση Βόλστομ. Ε, τα συμπεράσματα είναι ορθά και ισορροπημένα και η υιοθέτηση αυτών θα αποτελούσε ένα βήμα προς την ειρήνη. Αυτή την ε, ελπίδα έχουν έχουμε όλοι και οι μεγάλες δυνάμεις όμως δεν επιδεικνύουν θάρρος και πίστη προς τις δικές τους αξίες. Το να οργανώνει κανείς αποστολές παρακολούθησης εκλογικής δεν αρκεί όταν στη συνέχεια δεν γίνονται δεκτά τα αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και να έχουμε μια συνολική προσέγγιση για τα θέματα αυτά. Το Συμβούλιο θα έπρεπε να υιοθετήσει σύντομα ένα πρόγραμμα δράσης προς την κατεύθυνση αυτή με μια πραγματική στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να επιβληθεί σε όλα τα επίπεδα της Ένωσης με τις προτεραιότητες που είναι οι δικές μας, ούτως ώστε να ενταχθούν με τρόπο συγκεκριμένο στο σύνολο των μέσων μας εξωτερική πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτυξιακή πολιτική ε, παρακολούθηση στις τρίτες χώρες, τι γίνεται μετά, μετά την παρακολούθηση των εκλογών για να τηρηθεί ο πλουραλισμός, ο δημοκρατικός και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ποιες είναι οι απαιτήσει μας όσον αφορά την ε, θέσπιση μιας ανεξάρτητης ε, δικαιοσύνης και ε, διαφανών θεσμών απέναντι στους πολίτες. Η ασάφεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις πολιτικές μας είναι κάτι το αντιπαραγωγικό ε, πρέπει να διευκρινίσουμε τα πράγματα αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να λάβει υπόψη πιο σοβαρά ε, σε διεθνές επίπεδο τα ανθρώπινα δικαιώματα. μέρους του Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουλευτά. Η έννοια φτώχεια ορίζεται με πάρα πολλές ε, ερμηνείες. Ε, μία από αυτές είναι η έλλειψη της ασφάλειας. Η εξέλιξη λοιπόν αναχαιτίζεται χωρίς την ελευθερία και χωρίς την ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Άρα δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει και ανάπτυξη χωρί, χωρίς ειρήνη. Για να υπάρξει αυτό προϋποτίθεται ότι υπάρχει και απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά λοιπόν είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τη δημοκρατία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με στήριξε στην εργασία μου ως ε, βουλευτής ε, μετά από 7 χρόνια σε αυτό το αξίωμα ξέρω ε, πολύ καλά το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για την προώθηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία που ανελήφθη από την Τσεχική Προεδρία συζητήθηκε ήδη με την αδελφό μου, κυρία Γκούναλα Χάλστρομ, και η πρωτοβουλία αυτή θεωρεί ότι η δημοκρατία αποτελεί ε, στοιχείο κλειδί στη συνεργασία τόσο με τις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφαλείας. Εμείς όμως θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Θέλουμε να είμαστε ο παίκτη με 27 μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σημαντικός παράγοντας στην οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές της σχέσεις. Και ελπίζουμε η πρωτοβουλία μας θα αποτελήσει έναυσμα ε, για συνεργασία με όλες τις χώρες του κόσμου. Όμως θέλουμε να έχουμε και μια ρεαλιστική πρωτοβουλία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική χρήση όλων εκείνων των μέσων που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμών. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά. Η εμπειρία μας από άλλες καταστάσεις στον ε, τομέα της ε, εξωτερικής πολιτικής. Η εμπειρία μας λοιπόν αυτή όπως και η προσχώρηση των ε, τελευταίων χωρών αλλά και οι σχέσεις μας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας όλο αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις και διορθώσεις. Μπορούμε να κάνουμε πολλά και καλύτερα. Χρειαζόμαστε ένα πολιτικό εργαλείο, πλαίσιο και επιμέρους μέτρα τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά, θα ε, συντονίζονται μεταξύ τους και θα συμπληρώνονται. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και έτσι θα βελτιωθεί και η αξιοπιστία των εργασιών μας. Νέα λοιπόν μέσα είναι απολύτως απαραίτητα. Αν δεν τα βρούμε αυτά, τότε θα βλάψουμε την εξέλιξη. Πώς θα προχωρήσουμε τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και σωστά και ήδη έχει σημειωθεί επιτυχία. Παραδείγματο χάρη η στράτευσή μας στα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί αυτή ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ο πρώτος και ο τρίτος πυλώνας είναι επίσης ένα παράδειγμα ότι έχουμε δημιουργήσει ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας και αυτό αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για την οικοδόμηση της δημοκρατίας. Με αυτές τις προσπάθειες ε, σφυριλατούμε και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε βέβαια και μετριοπαθείς γιατί οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Γνωρίζω πολύ καλά ότι επικρατεί ανησυχία για το ότι στην αναπτυξιακή εργασία εισάγονται νέοι θεσμοί. Όμως μιλάμε και εμείς ε, για ανθρώπινα δικαιώματα και για δημοκρατία με τους ε, εταίρους μας. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που διαφαίνονται αυτή τη στιγμή. Εμείς θα οικοδομήσουμε ε, σε αυτά που έχει επιτύχει η Τσεχική ε, Προεδρία, η οποία οργάνωσε και ένα συνέδριο με αντικείμενο τη δημοκρατία. Ε, θέλουμε να υπάρχει ένα Ινστιτούτο για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και εδώ έχουμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η διαδικασία έχει προχωρήσει με συγκεκριμένα μέτρα, αρκετά ικανοποιητικά. Τα θέματα της δημοκρατίας συνδέονται με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι εργασίες προχωρούν και παράλληλα και από κοινού. Εμείς επιδιώκουμε ήδη τον Νοέμβρη να εγκριθούν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί, που αφορούν βέβαια και συγκεκριμένες μεμονωμένες χώρες. Και ε, οι προτάσεις αυτές ε, συνοδεύονται και με ενδελεχή ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στις διάφορες χώρες. Ε, η συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε διαβουλεύσεις, σε διάλογο, η οικοδόμηση της δημοκρατίας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα θέμα αυτό καθεαυτό και να υπάρχει επ' αυτού καλύτερος συντονισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει τις ε, εκλογικές διαδικασίες σε όλες τις χώρες και εμείς ανησυχούμε για το ότι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας να παρακολουθεί κανείς ε, τις εξελίξεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντάξει, να παρακολουθεί κανείς τις εκλογές, αλλά όχι μόνο αυτές, να ε, παρακολουθεί κανείς και το τι συμβαίνει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ανάμεσα στις εκλογές το, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πολύ σημαντικός σε όλη αυτή τη διαδικασία της οικοδόμησης δημοκρατίας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις ευκαιρίες. Ελπίζουμε η συνθήκη της Λισαβόνας να τεθεί σύντομα σε ισχύ και τούτο σημαίνει ότι θα έχουμε μια αποτελεσματικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη θα εμφανίζεται ως ε, ισχυρότερος πρωταγωνιστής στα πολιτικά δρόμενα και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα τύχει καλύτερου συντονισμού και οι εργασίες ε, της Κομισιόν και του Συμβουλίου θα συντονίζονται στο μέλλον καλύτερα. Εμείς λοιπόν ελπίζουμε μέσα από αυτή την ατραπό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προάγει με καλύτερα και αποτελεσματικότερα μέσα τις εξελίξει σε άλλα μέρη του κόσμου. Ένα δημοκρατικό κράτος το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των πολιτών του προκαλεί έλλειμμα δημοκρατίας. Και έτσι λοιπόν η οποιαδήποτε κυβέρνηση χάνει σε νομιμότητα και υποστήριξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πίεση που ασκούν ε, σε νομοθετικό επίπεδο, συνάπτοντας σχέσεις ε, με άλλα κοινοβούλια, στο ρόλο τους ε, ως παρατηρητές εκλογών, στο ρόλο τους ως συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο και ελπίζω να το διαφυλάξει για μεγάλο κόμμα χρονικό διάστημα. Ε, Δεν βλέπω τον κύριο Σαλαφράγκα στην αίθουσα και εκ μέρου ε, των σοσιαλιστών και των ε, δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μιλήσει η κυρία Ντεκάιζερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πώς να φέρουμε τη δημοκρατία σε μια χώρα στηριζόμενοι στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, ενισχύοντάς τη, καταπολεμώντας τον αποκλεισμό, την ένδια, ε, αφήνοντας τις γυναίκες να χειραφετηθούν. Με τα τάγκ και τις, και τις βόμβες δεν γίνεται, παρόλο που ορισμένοι το προσπάθησαν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μια ήπια δύναμη, soft power, όπως λέμε και θα πρέπει στην πρωτοβουλία Δημοκρατία Θεμόλη Δικαιώματα να δώσουμε περισσότερα δικαιώματα. Είναι εύθραυστο το βρέφος αυτό που βρίσκεται ακόμα σε εμβριακό στάδιο. Πρέπει να το ενισχύσουμε. Η μη ε, της επίσης. Ε, και είναι λίγη η πόρη αυτό της ε, πρωτοβουλίας ε, που κυρίως αφορούν τις αποστολές. Αποστολές που έχουν τεράστια σημασία διότι ήδη έδωσαν καρπούς αλλά για τις οποίες το Κοινοβούλιο ζητεί περισσότερα χρήματα, περισσότερη παρακολούθηση ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και πολύ α, περισσότερη πολιτική υποστήριξη. Συμφωνώ πλήρως με την κυρία Ζολή από τις αποστολές, σε σχέση με αυτό που είπε για από τις αποστολές μας. Δεν είναι λογικό να μην υποστηρίζουμε και μετά τις εκλογές ε, τις αναφιόμενες δημοκρατίες δεν πρέπει να βλέπουμε κοντόφθαλμα τα πράγματα. Είναι κάτι που η υπηρεσία των εξωτερικών σχέσεων βεβαίω θα συμπεριλάβει το δίχω άλλο στι μελλοντικέ του λειτουργίε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριο Γκέρεντ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει δημοκρατία χωρί ελευθερία. Όχι. Υπάρχει δημοκρατία χωρί δικαιώματα ή χωρί δίκαιο. Όχι. ένα σουφός Μπουρκιναβέζος είπε ότι αυτός που ζει στην απόλυτη ένδια δεν έχει ελευθερία, διότι δεν μπορεί να επιλέξει. Η ένδια άρα είναι συνώνυμο της στέρηση ελευθερίας. Ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στοιχεία μεταξύ τους και δεν αποτελεί καμία έκπληξη που αναφέρονται και οι τρεις αυτές έννοιες, τα κείμενα που μας συνδέουν με τις τρίτες χώρες, σύμβαση Κοτονού, ας πούμε, που έχει μία ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες ΑΚΕ. Η προώθηση της δημοκρατίας άρα θέτει θέματα ουσίας και αποτελεί την λεγόμενη ευφυή ύπαρξη προϋποθέσεων για τη χορήγηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Οι εταιρικέ σχέσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των τρίτων χωρών δεν μπορούν να το αγνοήσουν αυτό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρί αποφασιστικότητα, αλλά δεν μπορούμε να, να προχωρήσουμε και χωρί υπομονή. Χρειάζεται λοιπόν ο υπομονή με πολλέ από τι χώρε που βρίσκονται στο δρόμο της, ε, του εκδημοκρατισμού και πρέπει να συνοδεύσουμε αυτή τη διαδικασία χάρη σε μια στρατηγική που θα περιλαμβάνει μέτρα κατά της ένδυας, της κωδικοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισχύω των βασικών ελευθεριών και το κράτο δικαίου. Ακούσαμε όλες ε, τις ε, κριτικές που ακούστηκαν εναντί αυτή τη πολιτική, πολλές από τι οποίε συμμερίζομαι, αλλά αυτό το οποίο έχουμε κτίσει στο παρελθόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να το οικοδόμουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εκδημοκρατισμός είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει και με το σεβασμό των δικαιωμάτων και με διαχείριση τη εξουσία, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη του σκοπού εξωτερική πολιτική και θα πρέπει να συντονιστούμε για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο το, αυτό το οποίο έγινε και από το ότι υπήρξε συνένεση πανευρωπαϊκά και συγχαρητήρια στη Σουηδική Προεδρία για αυτή την πρωτοβουλία σχετικά με την καταπολέμηση τη φτώχεια. Πρόεδρε, πιστεύω κρατά ότι ο δημοκρατισμό θα πρέπει να καλύψει όλε τι πολιτικέ λόγε ενό για τι τρίτε χώρε. Και ε, επίση καταδικάζω τους ε, συντηρητικούς διότι είναι κατά τις διατάξεις που 10 στο κείμενό μας γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουν α, άλλα να λέει η, Ευρώπη και, και, και άλλα να κάνει όταν δεν τη βολεύουν αυτά που έχει πει. Τέλος, όπως είπε και η κυρία Υπουργό, η οικοδόμηση της δημοκρατίας είναι πολύ περισσότερο από το να κάνουμε εκλογέ. Είναι ε, ε, το χτίσμα μιας πλουραλιστικής κοινωνίας και γι' αυτό και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις μη κυβερνικές οργανώσεις, να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών, θα πρέπει οι περιθωριοποιημένοι να εμπλακούν, να συνεργαστούμε με τους, ε, τις και τους φορείς τους, να ενδυναμώσουν τα πολιτικά κόμματα ε, για το ε, κοινοβούλιο και τελικά δημοκρατία σημαίνει να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών να αναδείχθει. Κύριε Χάρη, σας ευχαριστούμε το πρώτος και τώρα. Η διαδικασία κάτσε και βλέπω εκεί την κυρία να δει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με την ε, οικοδόμηση τη Δημοκρατία το τι γίνεται προ Ανατολά με του γειτονέ μα. διότι τα τελευταία χρόνια είχαμε εκεί μια, σταθερότητα ή και ένα πισωγύρισμα όσον αφορά την, τον εκδημοκρατισμό αυτών των χωρών. Ε, τα γεγονότα στην ε, Μολδαβία και στην Γεωργία μα ενισχύουν πάρα πολύ διότι η σπονδική στήριξη κάθε δημοκρατική χώρα πέραν τη λειτουργία είναι το να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία τη κοινωνία των πολιτών. Κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά και απουσιάζει σε όλε τι ε, χώρε προ προσανατολά τη ε, Ένωση. Με συγχαρητήρια στην Σουηδία γιατί βοήθησε να υπάρχει πολιτική γειτονία, διότι με αυτή την πολιτική μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά του γείτονε μα προ Ανατολά από πολλέ απόψει. Αυτή η εταιρική σχέση. Θα πρέπει όμως να δημιουργήσει αληθή αυθεντικά κίνητρα γιατί πρόκειται για μια μακρά υπόδειγμα διαδικασία ούτω ώστε να κάνουμε μεταρρυθμίσει σε αυτέ τι χώρε. Οπότε έχω μια ερώτηση συμπληρωματική. Τι πρεσβεύει σχετικά με αυτό το συμβούλιο, Τι έχει κατά να κάνει. Και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία και σε εκείνη την περιοχή του κόσμου αλλά και σε άλλες που έχουν τέτοια προβλήματα θα ενδυναμωθεί. Κυρία Χαουτάλα, έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω, να ρωτήσω κάτι την κυρία Μάλστρομ. Νομίζω ότι μια από τις αδυναμίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις προσπάθειες μας υπέρ της δημοκρατίας έχει δύο στοιχεία. Αφενός τα κράτη-μέλη έχουν στόχους που είναι καμιά φορά ε, αντιφατικοί, έρχονται σε αντίθεση παραδείγματο χάρη η απαγόρευση εξαγωγής όπλων σε σχέση με το Ουσμπεκιστάν και πώς με τον τρόπο αυτό θα ήταν δυνατόν να έχουμε μια κοινή πολιτική. Δεύτερον, το Ουσμπεκιστάν δίνει το παράδειγμα μιας χώρας που λέει εσείς Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχετε μαθήματα να μας δώσετε ως προς την δημοκρατία διότι έχετε τα δικά σας κενά και τις δικές σας ελλείψεις. Πώς θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από αυτήν τη διγλωσία διότι αφενός θέλουμε να διδάξουμε τους άλλους αλλά δεν κάνουμε αυτά που απαιτούνται ε, ε, στο δικό μας το σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την ε, δημοκρατία. Ε, ποια οργάνωση μίλησε για αυτή τη διγλωσία. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αν όχι, θα ζητήσω από την κυρία Μάλστρομ να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη δημοκρατία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Κυρίως τώρα, με μεσούσεις ε, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε αυτή τη διάσταση του θέματος. Πάρα πολλά αναπτυσσόμενα κράτη πλήττονται από την κρίση. Η ύφεση προκαλεί κοινωνικές αναταραχές, ε, δυσαρέσκεια ε, και χωρίς δημοκρατικούς θεσμούς τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πολύ δυσάρεστα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν καλοί δημοκρατικοί θεσμοί και μια ισχυρή ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Ως προς την ε, ε, συνεργασία με τις ανατολικές χώρες, αυτό το εργαλείο που υπάρχει είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Ε, για το Δεκέμβρη προβλέπουμε μια σχετική συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών και στις αρχές του επόμενου έτους θα ασχοληθούμε εντατικά με το θέμα αυτό. Διότι ε, βρισκόμαστε σε απόλυτη γυτνίαση με τις χώρες αυτές. Όσον αφορά την ερώτησή σας για το Ουσμπεκιστάν, βεβαίως αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουσμπεκιστάν επουδενή δεν μας ικανοποιεί και σήμερα δεν υπάρχει πλέον ομοφωνία στο Συμβούλιο. Όμως ε, όλοι μας ε, επιδιώκουμε τον ίδιο στόχο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον με το να ε, ασχολούμεθα συνεχώς με το θέμα αυτό και με το να ορίσουμε τι είδους σχέσεις θέλουμε να έχουμε με το Ουσμπεκιστάν υπάρχουν ενδεχομένως άλλα μέσα που θα μπορούσαν να κρυθούν ε, περισσότερο αποτελεσματικά ε, από το εμπάργο όπλων. Γιατί αυτό το εμπάργο είναι περισσότερο ένα συμβολικό μέτρο. Για να καταλήξουμε όμως σε άλλα μέτρα χρειαζόμαστε ομοφωνία η οποία δεν υφίσταται σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμφανίζεται αξιόπιστη. Γιατί οποτεδήποτε μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, τούτο σημαίνει ότι πρέπει και στο εσωτερικό μας να είμαστε ισχυροί. Βεβαίως και υπάρχουν υπάρχουν ελλείψεις, κενά και για το λόγο αυτό οφείλουμε ακαταπώνητα να προσπαθούμε να είμαστε αξιόπιστοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση και για το ψήφισμα το οποίο βρίσκω και εξαιρετικό. Ψήφισμα το οποίο αντικατοπτρίζει απόλυτα τις απόψεις της Σουηδικής Προεδρίας και ελπίζουμε το Νοέμβρη να μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε για το θέμα αυτό και χαιρόμαστε για περαιτέρω συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό.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 Και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα τη μέσης διάταξη που είναι οι ερωτήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.